Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόταση. Περνάμε στις ψηφοφορίες τώρα. Η ε, γραπτή δήλωση των κυρίων Μέγερ, για την επιστροφή της τους στις ε, κατοίκους της έχει υπογραφεί από την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζασάντα για ένα λεπτό. Ένας από τους υπογράφοντες του αιτήματο. Κύριε Ζασάντα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι και συνάδελφοι. Υπάρχουν ορισμένες ε, περιοχές, ορισμένα μέρη στην Ευρώπη και υπάρχει μια συγκεκριμένη πόλη στην Κύπρο, στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι περιφραγμένη με ε, σειρματόπλεγμα. Έχουμε ε, χιλιάδες, εκατοντάδες και σπίτια καταλελειμμένα, εκκλησίες, σχολεία, ε, γήπεδα. Οι κάτοικοι της πόλης αυτής περιμένουν τη μέρα που θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ε, στα παιδικά τους σπίτια. Για να υλοποιηθεί αυτό το όνειρό τους, για να γίνει πραγματικότητα, χρειάζεται σημαντική βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και για τη βοήθεια αυτή ε, και προσωπικά και Εξ ονόματος των υπογραφών της ε, γραπτής δήλωσης υπαριθμών 42 και ιδιαίτερα εξ ονόματος ε, των ε, κατοίκων της αμοχώς του, των παιδιών και των εγγονών τους θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί γνωρίζω ότι με την ανακοίνωση αυτή θα δοθεί έναυσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τα κράτη-μέλη στον ΟΗΕ και ιδιαίτερα στην τουρκική κυβέρνηση για να ενισχυθεί η συνεργασία και να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ θερμά.